Τώρα, προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Καταρχήν, έκθεση Winkler. Ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Did Ψηφίσατε. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Μια scheda το mio posto, Μια μια scheda. Approved with the large majority. Εγκρίνεται με ευρεία πλειοψηφία. Έκθεση Ντεκάστρο, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ναι. Πέρας. Εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Συγχαίρω τον κύριο Ντεκάστρο και τον κύριο Βίγκλερ. Έκθεση Χάτων εισηγητής έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή ψηφίζεται σήμερα γιατί είχαμε σημαντική καθυστέρηση για το πότε καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και αυτό δεν προξενεί εκπλήξη καθώς είχαμε γύρω στις 2.600 τροπολογίες που κατατέθηκαν από συναδέλφους. Αλλά η έκθεσή μου είχε παρουσιαστεί ως καθαρά τεχνικό ζήτημα αλλά υπάρχουν νομίζω κάποια ουσιαστικά μηνύματα. Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Αλληλείας κάτι το οποίο είναι και αυτό ασύνηθες και σκοπεύει να διασφαλίσουμε πως ε, το καστό πρόσβασης ε, στα 12 μίλια θα συνεχίσει να υφίσταται και βεβαίως ε, με την νέα αλλιευτική πολιτική. Εάν δεν εγκρίναμε αυτή την αλλαγή θα εξέπνεε στο τέλος του έτους η πρόσβαση στα 12 μίλια και αυτό θα ήταν βεβαίως αδιανόητο και ανεπίτρεπτο. Η ζώνη των 12 μιλίων ήταν χαρακτηριστικό της κοινής αλληλευτικής πολιτικής από τον αρχικό κανονισμό το 1983 και τώρα θα ισχύσει για άλλα 10 έτη. Η παράταση αυτή δηλαδή θα ισχύσει μέχρι το 2014 πρώτα και μετά θα δούμε ποια θα είναι η νέα κοινή αλληλευτική πολιτική. Αλλά ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεχτεί πως η διαχείριση των αλληλευμάτων εντός της ζώνης των 12 μιλίων ήταν συνολικά επιτυχής. Οπότε, αντλώντας διδάγματα από αυτό, κάτω σημαίνει πως τα κράτη τα ίδια ε, ήταν ε, επιτυχή στην διαχείριση αυτή σε συνδυασμό με την αποτυχία της κοινή αλλιευτικής πολιτικής νομίζω πως μπορούν να μας οδηγήσουν στο να επεκτείνουμε τα 12 μίλια και χρονικά και τοπικά. Αλλά αυτό είναι ζήτημα μιας άλλης έκθεσης την οποία αναμένω. Σας ευχαριστώ. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Παρακαλώ. Θα σας περιμένουμε. Ωραία, πέρας. Ομόφωνα. Συγχαίρω τον εισηγητή. Έκθεση Μορέιρα. Κύριε Μορέιρα, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομος. Έχω κάτι σημαντικό να σας πω. Πρώτα απ' όλα, ως εισηγητής, σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε αυτή τη συμφωνία γιατί είναι μια καλή συμφωνία και πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα για μελλοντικέ συμφωνίες στο θέμα αυτό και ελπίζω να έχουμε ομοφωνία. Όμως, εγκρίνοντας αυτή την συμφωνία δεν ψηφίζουμε ούτε αποδεχόμαστε την απόφαση του Συμβουλίου επί του θέματος γιατί υπάρχει μια διάταξη η οποία ορίζει ένα μηχανισμό επιτροπολογίας μέσω μιας διαδικασίας εξέτασης που θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να ελέγχει τις αποφάσεις της Κομισιόν όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Κατά την άποψή μου, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να δεχτεί το Συμβούλιο να αποφασίζει μόνο μερός για κάτι το οποίο εξορισμού θα πρέπει να είναι στην συναπόφαση. Πόσο μάλλον να δεχτούμε να γίνεται κατάχρηση της διαδικασίας της επιτροπολογίας από το Συμβούλιο έτσι ώστε μονομερός και ε, ε, και μονομερός να ελέγχει το Συμβούλιο της Αποφάσης Κομισιών. Οπότε πρέπει να είναι σαφές πως δεν εγκρίνουμε το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου επί του θέματος και αν παραμε, παραμείνει το σχέδιο το ίδιο, κάτι το οποίο ελπίζω ότι δεν θα γίνει, δεν θα επιτρέψουμε να θεωρηθεί προηγούμενο για μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες. Δυστυχώς δεν είναι εδώ το Συμβούλιο, αλλά είμαι σίγουρος πως το μήνυμά μου θα φτάσει. Σας ευχαριστώ. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση Ντίβα. Κύριε Ντίβα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο για το ότι επέτρεψαν να περάσει τόσο γρήγορα η έκθεση. 15.000 άνθρωποι θα πεθάνουν από την πείνα σήμερα. Για να καταλάβετε, πρόκειται για το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο ε, και το προσωπικό τους και το 1 τρίτο της Κομισιόν. Η συνολική ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να διπλασιαστεί να φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους μετά να φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους και θα πρέπει η παραγωγή των τροφίμων να διπλασιαστεί. Η φυστάμενη συμφωνία διατροφικής βοήθειας δεν επαρκεί. Η νέα συμφωνία, την οποία θα ψηφίσουμε σήμερα, θα εισαγάγει νέες μορφές ε, βοήθειας. Τοπική παραγωγή με τοπικές αγορές, ε, διατροφική βοήθεια χωρίς όρους, ε, κουπόνια σε αγρότες με τα οποία μπορούν να αγοράζουν, τα οποία μπορούν να εξεργειώνουν σε χρήματα και τροφή και βοήθεια σε αναψώμενε χώρες. Σας ευχαριστώ όλους που εργαστήκατε τόσο σκληρά για να περάσει αυτή η έκθεση και για το ότι προσπαθείτε να σώσετε τόσες ζωές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση Bauer. Ο εισηγητής ζητάει το λόγο. Ε, η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία γιατί συζητήθηκε στην Ολομέλεια η έκθεση. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η προτινόμενη οδηγία σκοπεύει να αντικαταστήσει την απόφαση του 1995 όσον αφορά την προξενική προστασία πολιτών της Ένωσης από διπλωματικές και προξενικές αρχές δεδομένου του νομικού πλαισίου της συνθήκης της Λισαβόνας το άρθρο 23 της Συνθήκης Λισαβόνας πάνω στο οποίο βασίζεται η ε, πρόταση προβλέπει πως κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικράτεια τρίτης χώρας στην οποία δεν εκπροσωπείται η χώρα του θα δικαιούται προστασίας από προξενικέ και διπλωματικές αρχές. Η πρόταση καλύπτει όχι μόνο καθημερινές καταστάσεις όπως απώλεια διαβατηρίου, ε, εγκλήματα, ατυχήματα αλλά και θάνατο, αλλά και καταστάσεις κρίσης όπου ίσως χρειαστούν βοήθεια οι πολίτες της Ένωσης. Ενώ στις καθημερινές προξενικές υποθέσεις οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν βοήθεια σε οποιοδήποτε προξενείο πρεσβεία. Οι καταστάσει κρίση όμως είναι διαφορετικέ. Η Επιτροπή συμφώνησε σχεδόν σχεδόν ομόφωνα πως ε, δεν θα πρέπει να επομίζεται κάποιο κράτος μέλος το βάρος αυτό, οπότε θα πρέπει το βάρος αυτό να βγαίνει στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει ότι περισσότερη Ευρώπη δεν σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία, αλλά περισσότερη βοήθεια για τους Ευρωπαίους πολίτες όταν το έχουν ανάγκη, περισσότερη προστασία για αυτούς οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται σε τρίτες χώρες που βρίσκονται σε καταστάσεις ε, επικίνδυνες οι καταστάσεις κρίσης. Τέλος, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις ε, εισηγητές για την προσπάθειά τους και να ε, ζητήσω από όλους τους συναδέλφους να ε, το στηρίξουν. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση μπάστος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συγχαρητήρια. Έκθεση Μπόουλς Τι θέλετε. Μυστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. κύριος Καμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως είναι απαράδεκτο να ψηφίζουμε υπέρ ή κατά ενός ανθρώπου. Είναι μυστική ψηφοφορία, αλλά το, το όνομά του δεν είναι μυστικό. Δεν είναι κοινοβουλευτική αυτή η διαδικασία. Το όνομα δε του ανθρώπου δεν εμφανίστηκε καν στην οθόνη. Gli uffici mi dicono che abbiamo rispettato pienamente la procedura per cui il voto è valido. Μου λένε ότι τηρήσαμε τη διαδικασία, ισχύει η ψήφος και προχωρούμε. Έκθεση Μορέια. Amendment 1. Τροπολογία υπάρχει μόνο ένα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. ψηφίσουμε την έκθεση στο σύνολό της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η έκθεση ονομαστική αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται συγχαρητήρια Επόμενη έκθεση, επόμενο θέμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι. Έκθεση Σνίμπερ Γιάστραμ. Παράγραφος 3, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 23. Πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την παράγραφο 36. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα έχει το λόγο. Α, δεν ζητήσατε το λόγο. Με συγχωρείτε. Α, ναι, ναι. Έχετε το λόγο. Η τροπολογία μετά το child prostitution θα θέλαμε να λέει ενώ προστατεύει τις γυναίκες έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες και υπηρεσίες ε, αναπαραγωγής και προστασίας. Νομίζω κανείς δεν αντιτίθεται. Εντάξει, λυπάμαι. Κύριε Κόρτες Λάστρα, δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί αυτή η προφορική. 144. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές Ελέγχουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. The Πέρας. Εγκρίνεται. 147. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος, εντάξει, ελέγχουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 148. 148. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Εντάξει. Αρχίζει η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν κάνουμε αυτή τη σημαντική ψηφοφορία, θέλω να σκεφτούμε τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων από την άλλη πλευρά που ορθώθηκαν για να στερήσουν από τις γυναίκες τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Εντάξει. Το λόγο θα το δώσω μόνο στον κύριο Μίτσελ και μετά κανένας άλλος. Ο λόγος για τον οποίο εγώ σηκώθηκα είναι ότι 200 εκατομμύρια γυναίκες λείπουν από τον παγκόσμιο πληθυσμό λόγω των αμβλώσεων που γίνεται υπέρ με βάση το φύλλο. Θα πρέπει να, να... Ε, επιτρέπ... να μην επιτρέψουμε να χάνονται γυναίκες επειδή είναι γυναίκες. Okay. Roll call. Ονομαστική ψηφοφορία έναρξη. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Συγχαίρω τον εισηγητή. Καλή σας όρεξη. Παλιά το μόνο. Please, please, Αγαπητοί συνάδελφοι. Εν τω μεταξύ λειτουργήσε η μηχανή μου, μετά σταμάτησε, μετά ξαναπήρε μπρο. Είχα πρόβλημα δηλαδή με το μηχάνημά μου στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay, we inform the... Μάλιστα θα ενημερώσουμε τις υπηρεσίες. Τώρα και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου.